Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε όλους παρόντες όσοι πρέπει να είναι παρόντες. Λοιπόν, προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο Οριθέτηση Μειονεκτικών Περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ΚΑΠ. Η κυρία Κόστινγκερ έχει πρώτη το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο που εμφανίστηκε. Πρόκειται για πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα ε, που έχει μεγάλη, και έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε τη συζήτηση αυτή απόψε μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει νέα αξιολόγηση των ε, μειονεκτικών περιοχών το Μάιο του 2001 είχαμε κάνει μια έκθεση και εκφράσαμε επιφυλάξει για το νέο μοντέλο. Η πρόταση προβλέπει ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 8 ε, ε, βιοφυσικά κριτήρια για εδαφολογικά, κλιματικά κριτήρια για να οριστούν οι μειονεκτικές περιοχές. Αυτό είναι μοιραίο για ορισμένες περιοχές. Συνάδελφοι, για τη διερμηνία μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ. Τα νέα κριτήρια σημαίνουν ανακατανομές στις περιοχές. Αυτό το ξέρουμε για κάποια κράτη-μέλη. Οι λεπτομερείς οι υπολογισμοί και οι προσωμιώσεις δεν υπάρχουν όμως για περαιτέρω διαπραγμάτευση της κοινή αγροτικής πολιτικής όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει ως συνομοθέτης θα πρέπει όλα τα στοιχεία να τα έχουμε επιτάπητος. Εμείς δεν θέλουμε ευαίσθητες περιοχές που προφανώς πλήττονται από ε, φυσικές ε, μειονεξίες να φύγουν από το χάρτη. Τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο και πότε θα λάβουμε όλες τις προσωμιώσεις. Θα πρέπει το Συμβούλιο να φροντίσει ώστε το Κοινοβούλιο ε, να μην υστερήσει σε ενημέρωση στη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να βρεθούν καλές λύσεις για τους αγρότες και τις αγρότησες. Μέχρι να δοθούν όλα τα δεδομένα επιφυλασσόμεθα ε, να αποκλείσουμε από τη μεταρρύθμιση το θέμα των μειονεκτικών περιοχών. Επίσης ε, πιστεύω ότι οι ανησυχίες μας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, προγράμματα που να επιτρέπουν τη συνέχιση των εργασιών και τη δημιουργία εισοδήματο από τις εκμεταλλεύσεις ε, και όχι να του θερήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε μια δέσμη κριτηρίων για τη διατήρηση των εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική απόδοση και αυτό για όλες τις, ισχύει για όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτό το πλαίσιο. Περιμένουμε ε, από εσά ε, μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ε, για δύο λεπτά ο κύριος Καπούλα Σάντος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, το να εξασφαλίζεται η αγροτική δραστηριότητα στην Ήπεθρο είναι κάτι που αξίζει την έγκρισή μας. Θέλουμε να μείνει βιοπικιλομορφία, θέλουμε να αποφύγουμε τις δασικές πυρκαγιές, καλύτερη διαχείριση των υδάτων, καλύτερη προστασία των εδαφών. Όμως, γι' αυτό συζητούμε σήμερα. Αυτό που συζητούμε σήμερα ε, είναι πρακτικής φύσεως. Εμείς που θέλουμε να ετοιμάσουμε την έκθεση για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να αποφασίσουμε και να νομοθετήσουμε χωρίς να έχουμε πληροφορίες όσον αφορά τις πραγματικές συνέπειες και τα κριτήρια τα πραγματικά, τα τοπικά. Το Συμβούλιο θα πρέπει να μας ενημερώσει. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε ήδη να διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τις πραγματικές συνέπειες των νέων κριτηρίων στα κράτη-μέλη. Το ερώτημα που έχω να θέσω προς το Συμβούλιο είναι το εξή. Μπορείτε να μου πείτε αν το Συμβούλιο μπορεί να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες. Και αν ναι, πότε. Θα ήθελα να επενθυμίσω επίσης στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και ένα μήνα εδώ σε ένα μήνα, σε ένα μήνα μάλλον, οι συγγητές θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους. Αν μπορούμε και να διαθέτουμε αυτές τις πληροφορίες, θα είναι καλό. Διαφορετικά δεν μπορούμε να νομοθετούμε υπεύθυνα χωρίς πληροφορίες. Εφόσον τα Συμβούλια και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα, θα ήθελα πραγματικά το Συμβούλιο να μας πει ξεκάθαρα, ειλικρινά, εάν θα μπορέσει να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και πότε. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μας, ε, για τη δουλειά μας ως νομοθέτες. Ευχαριστώ. Επόμενος ο μιλητής για δύο λεπτά ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό το πρόγραμμα, κυρίως στη Βόρεια Ιρλανδία. 70% της γεωργίας ε, ε, ε, είναι σε μη πολύ ευνοϊκή περιοχή και οι πληρωμές που δέχονται οι υγρότε από το σχήμα είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τη ζωή του και κυρίω διότι είναι μόνο με μερική απασχόληση Γεωργή. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε την υιοθέτηση του σχήματο και αλλαγή των κριτηρίων για περιορισμού του σχήματο του προγράμματο μεγάλη προσοχή. Οι προβλέψει διατείνονται ότι σύμφωνα στις παρούσε προτάσει. Πολλέ επιλέξιμε γέε του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι τώρα επιλέξιμε, θα χάσουν το καθεστώ αυτό. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια περίπου το 30% ε, γεών. Ε, κάποιες περιοχές μπορούν να χάσουν πλέον παραγωγικές γέες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο νέο σχήμα όμως. Περιοχές που ίσως να μην απαιτούν όμως τέτοιου είδους υποστήριξη. Και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έκανε σωστή αξιολόγηση νεπιών όσον αφορά την προτινόμενη κοινοποίηση. Θέλω να ισότιμε συνθήκε για όλα τα κρατη Αυτό απαιτεί αναγνώριση όλων των ειδών φυσικών περιορισμών που είναι επιζήμιοι για την αγροτική παραγωγή. Δάτω μας ευκαιρίες να πω το εξή. Μεγάλοι, πολλές βροχές, όπως στην περιοχή μου, μπορεί να εξίσου καταστροφικές για την καλλιέργεια, όπως η ξηρασία σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και γενική προσέγγιση δεν ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση για να διαφυλάξουμε την αποτελεσματικότητα του σχήματο που προτείνεται, θέλω ευρεία, ευέλικτη προσέγγιση. Το παρόν σχήμα λειτουργεί άριστα, πιστεύω. Και δεν θέλω να υπονομευτεί επουδενή. Διερωτώ με, ποιο καθοδηγεί την ΚΑΠ και τη μεταρρύθμιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ελεκτικό Συνέδριο τελικά. Φαίνεται το ελεκτικό συνέδριο επέκρινε κάθε κίνηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή την εβδομάδα όσον αφορά το πακέτο μεταρρύθμιση. Αν η μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίδραση του ελεκτικού συνεδρίου που θεωρεί μη δικαιολογημένε πληρωμέ, αν αυτό ισχύει και επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελεκτικού συνέδριου, σκανδαλώδε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, για δύο λεπτά ο κύριο Λάιον παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στην Σκοτία 85% είναι το επιλέξουμε οπότε και εμείς με αγωνία περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα νέα κριτήρια. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε πάρα πολύ θα αισθανθούσαν να είναι επιλέξιμοι όμως τελικά έγινε κάποια διόρθωση στα σχετικά δεδομένα και η Κομισιόν περιέλαβε και ε, την, την ξηρασία ή μη ξηρασία του εδάφους ως κριτήριο λήφθη αυτό υπόψη και έτσι ξανασχεδιάστηκε ο χάρτης Ιδίω αποκαταστάθηκαν διάφορες περιοχές στην Ανατολική ακτή. Και έτσι επομένως αποχαρακτηρίστηκαν ως ε, προνομιούχε κάποιε περιοχέ. Πάντω οπωσδήποτε έχουν υπάρξει σημαντικέ συνέπειε από αυτά τα μέτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα και στη Σκοτία, και όπω βλέπετε μπορεί να δει κανεί οποιοδήποτε τέτοιο χάρτη και ε, σε άλλε χώρε όπω είπαν οι συνάδελφοι. Οι χώρε αυτέ, οι κυβερνήσει, αναγκάζουν την Κομισιόν να μην κοινοποιεί τα σχεδιαστικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει επομένω να συμμορφωθούμε προς τα όσα ζητεί το ελεγκτικό συνέδριο. Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι επίτηδε αποκρύπτουν στοιχεία και συνάδελφοι μέλη τη Επιτροπής Γεωργίας. Θα πρέπει επομένω εμείς που είμαστε συνομοθέτες να έχουμε προσβασιμότητα, ισόρροπα στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Άρα, να μας αποκαλύψουν τα σχετικά στοιχεία αν θέλουν να προχωρήσει το θέμα της νομοθεσίας το συντομότερο δυνατόν. Όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να μας τα δίνετε. Να ξέρουμε ότι ξέρετε κι εσείς το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος Μπότσκοφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Ο Δανός Υπουργό Τροφίμων δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί απόψε, γι' αυτό εξ του Δανού Υπουργού και της Προεδρίας θα απαντήσω στις ερωτήσεις 70 και 71 για την οριοθέτηση των ε, μειονεκτικών περιοχών στα πλαίσιο της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής. Για να υπάρξει μια εποπτεία ε, μετά την εφαρμογή των 8 βιοφυσικών κριτηρίων για τις μειονεκτικές ε, περιοχές και την οριοθέτησή τους, η Κομισιόν ζήτησε από τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν χάρτες περιοχών. Πρόκειται για περιοχές ε, που θα δικαιούνται τις ενισχύσεις με βάση ε, προσωμιώσεις ε, για τη χρήση των κριτηρίων. Καταλαβαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να δει τους λεπτομερείς χάρτες και δυστυχώς αυτό ακόμη δεν μπόρεσε να γίνει. Το θέμα των νέων κριτηρίων για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών είναι τώρα τμήμα της μεταρρύθμισης κοινή αγροτικής πολιτικής. Όμως, ακόμη δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή των οκτώ βιοφυσικών κριτηρίων. Συμφωνώ με τους ερωτώντες ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια βασικά δεδομένα σχετικά με τις συνέπειες από τη χρήση και εφαρμογή βιοφυσικών κριτηρίων ε, για τις μειονεκτικές περιοχές και περιοχές με ισχυρούς περιορισμούς στη Γεωργία. Από ό,τι γνωρίζω όλα τα κράτη-μέλη έχουν δώσει προκαταρκτικές πληροφορίες και χάρτες δείχνοντας τι συνέπειες από τη χρήση των 8 βιοφυσικών κριτηρίων. Τα στοιχεία τα έστειλαν λοιπόν στην Επιτροπή. Αν και είναι προκαταρκτικά τα στοιχεία και οι πληροφορίες, είναι παρόλα αυτά χρησιμότατα, γιατί μπορούμε να δούμε τις συνέπειες από τη χρήση των νέων κριτηρίων. Και αυτό είναι σημαντικό και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο, γιατί έτσι θα κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Όμως το Συμβούλιο δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και τους χάρτες. Οι χάρτες ανήκουν στα κράτη-μέλη. Μπορεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να τα δουν όταν, μόνο και μόνο όταν τα κράτη-μέλη δώσουν εντολή για να παραδοθούν τα στοιχεία αυτά. Η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσει ή να διανύμει τις πληροφορίες αυτές χωρίς άδεια. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, τώρα 12 κράτη-μέλη έχουν ε, συμφωνήσει να δώσουν έγκριση στην Κομισιό να δώσει τα στοιχεία ε, για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών με βάση τα βιοφυσικά κριτήρια. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις 23 Απριλίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την προθυμία αυτή αντιλαμβανόμεθα ότι οι ερωτήσεις αφορούν το ζήτημα της πρόσβασης ε, και της διαφάνειας της ενημέρωσης. Στις 16 Απριλίου έγινε μια συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας και η Προεδρία ενεθάρρυνε τα κράτη-μέλη να επαναξιολογήσουν τη θέση τους και να δώσουν την άδεια ε, ούτως ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στη διαδικασία. Αυτά στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Μετά κάποια κράτη-μέλη θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν να δουν τις επιπτώσεις των προτινομένων αυτών βιοφυσικών κριτηρίων. Έτσι λοιπόν τώρα το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω τις ερωτήσεις αυτές. Προτείνω λοιπόν ερωτήσεις με λεπτομέρειες να τεθούν την επόμενη φορά που θα έρθει η Επίτροπος ε, στην Επιτροπή Γεωργίας 23 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Εξ του ΕΛ και δύο λεπτά, ο κύριος Ντόρφμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, με τη νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών ε, παίζεται ένα κακόγουστο αστείο και νομίζω ότι η απόψινή συζήτηση δεν θα βελτιώσει τα πράγματα. Ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν το ήξερα ομολογώ. Πριν από δύο χρόνια ε, είχε εγκριθεί η έκθεσή μου για το θέμα αυτό, είχαν γίνει πολλές προτάσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καμία πρόταση δεν συμπεριελήφθη στη μεταρρυθμιστική πρόταση της Κομισιόν, η οποία επιμένει στη δική της πορεία. Η νέα οριοθέτηση τι σημαίνει. Θα προσθεθούν κάποιες περιοχές και ποιες, θα αφαιρεθούν άλλες και ποιες. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Μπορεί να υπάρχει καλύτερη οριοθέτηση από την τωρινή κάποια κράτη-μέλη είναι 100% μειονεκτικές περιοχές, άρα είναι δυνατό να γίνει. Αλλά θα πρέπει να οριοθετήσουμε σωστά τις περιοχές και να όχι υπερβολικά πολλές. Γι' αυτό τα οχτώ κριτήρια που προτείνονται δεν είναι απόλυτα σωστά και αποτελεσματικά. Ε, επίσης, μέχρι τώρα δεν γνωρίζει τίποτα το Κοινοβούλιο για τις προσωμιώσει. Αυτό είναι παράλογο. Λέτε ότι οι χάρτε είναι, ιδιοκτησία, είναι στην κατοχή των κρατών μελών. Ε, αλλά ε, παρόλα αυτά κάποιοι υπουργοί ζητούν από το Κοινοβούλιο να τροποποιήσουν τα κριτήρια. Μα πώς θα το κάνουμε αυτό αν δεν ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά στην πράξη τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν, η ισχυρίζονται ότι το Κοινοβούλιο θα επιμείνει στην ε, οριοθέτηση ε, την παρούσα. Ε, αυτό είναι όμως παράλογο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ε, φροντίσετε για τη διαφάνεια και να επιτρέψετε στο Κοινοβούλιο να εργαστεί όπως πρέπει προς το συμφέρον του, και του, Συμβουλίου και της Κομισιόν και πάνω απ' όλα προς το συμφέρον των ίδιων των αγροτών. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για ένα λεπτό ο κύριος Δεκάστρο. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, τον γνωρίζει κανεί τα στοιχεία προσωμείωση των κρατών μελών όσον αφορά τα νευρικά στοιχεία που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τοπισμό των, των περιοχών είναι κάτι θεμελιώδε για το Κοινοβούλιο στα προνόμια που έχει ο συνομοθέτη. Λοιπόν, η αδιαφάνεια και ο δισταγμό διαβίβαση αυτών των στοιχείων στου εκπροσώπου των Ευρωπαίων πολιτών αποκαλύπτει μια τοποθέτηση των κρατών μελών και του Συμβουλίου που δεν γνωρίζουν ακόμα την επανάσταση τη δημοκρατική που προέρχεται από τις ηθήσεις Σαββόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συναποφασίζει σε θέματα γεωργικά και μαζί με το Συμβούλιο θέλουμε να τα ρυθμίσουμε την κοινή αγροτική πολιτική. Και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε λοιπόν καμία διαφορά μεταξύ των πληροφοριών που κατέχονται από τα δύο θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να είμαστε στις ίδιες συνθήκες με το Συμβούλιο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε πλήρη επιγνώση τα στοιχεία που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, υπενθυμίζω, που δεν μας δείχνουν τα στοιχεία όπου έχουν δηλωθεί από κάτι κράτη-μέλη και καποια κάτι κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν τελικά τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο. Καλούμε το Συμβούλιο να ζητήσει από τα κάτι μελη να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και να υπάρξει πλήρη συνεργασία υπό το φως μιας νέα θεσμικής πραγματικότητας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο. Επόμενος Εν ονόματι της Άντε για δύο λεπτά είναι η κυρία Ράιμερς. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμο συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ περίεργο που να συζητούμε εδώ και να αποφασίζουμε για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά δεν έχουμε τα απαραίτητα κριτήρια για την απόφαση. θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάποια κριτήρια να ορίσουμε τις απομακρυσμένες περιφέρειες ή τις μειονεκτικές ε, κλιματικές ε, συνθήκες ε, ε, και άλλα κριτήρια δεν λέω ότι δεν αξίζουν και δεν ισχύουν αλλά θα πρέπει να έχει λόγο το κοινοβούλιο χρειαζόμαστε χάρτες για τη νέα κατανομή των μειονεκτικών περιοχών για να δούμε αν έχουν νόημα τα 8 κριτήρια γιατί δεν μας τα δίνετε αυτά τα στοιχεία καχυποψία. Δεν ξέρω, θέλετε να είναι δυνατή η συναπόφαση στο Συμβούλιο. Εγώ είμαι αγρότησα και έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες επί της ουσίας αν με τα κριτήρια αυτά που δίνονται μπορεί να γίνει σωστά μια νέα κατανομή των περιφερειών. Γιατί υπάρχουν και άλλα κριτήρια που μπορεί να συνιστούν μειονεκτική θέση όπω είναι η έλλειψη υποδομή, η πρόσβαση στην αγορά εργασία και γενικά ιστορικέ ε, οικονομικέ συνθήκε. Επίση, διαφορετικό συνδυασμό των διαφόρων κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Έχει έρθει η ώρα για να μην πω ότι έχει περάσει και η ώρα από το να ε, ε, εξετάσουμε αντικειμενικά τα κριτήρια και τα στοιχεία. Αλλιώς θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που θέλουν να εξαιρεθούν αυτές οι μειονεκτικές περιοχές από την παρούσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Εξ ονόματος των Πρασίνων τώρα για ένα λεπτό και μισό το λόγο έχει ο κύριος Σμιθ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ, εγώ είμαι Σκοτσέζος και μιλώ και προς ένα ομόλογό μου από τη Βόρεια Ευρώπη και σοσιαδημοκράτη, αλλά νομίζω ότι σας έχει φέρει σε δινή θέση η κατάσταση. Ε, είναι απαράδεκτα αυτά και αδικαιολόγητα. Εμείς οι νομοθέτες πώς θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Στη Σκωτία 85% όπως ακούσαμε της επικράτειας είναι με ενεκτική περιοχή και για μας ε, και τους αγρότες μας είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είναι σημαντικό, είναι ψήστης της σημασίας, δεν είναι καθόλου έλασον ή δευτερεύον. Πώς παράγουμε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε ε, κάνει μοντέλα και χάνουμε 622 τετραγωνικά χιλιόμετρα με τα νέα κριτήρια σύμφωνα με τους υπολογισμούς και ε, κερδίζουμε 5.536. Ε, αυτά είναι ε, στοιχεία πάρα πολύ διαφανή και σωστά και αντικειμενικά όπως θέλει και η Σκοτσέζικη και θέλει και η Δανική κυβέρνηση να βλέπει τα ίδια. Αλλά δεν θα πρέπει με τυφλό τρόπο ε, και ενιαίο ε, ισοπεδωτικά να εφαρμόζω αυτά τα κριτήρια. Δεν είναι τρόπος αυτός λειτουργίας και εργασίας. Και θα παρακαλούσα να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους και το βλέπω στην έκθεση Dorfman. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αυτή την ε, ενημέρωση και ούτε πρόκειται να το κάνω. Πρέπει να μας ενημερώσετε εδώ και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Εξ ονόματος της ομάδας του των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για ένα λεπτό το λόγο είχε ο κ. Βοητσοκόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμμετέχω στα της χαρτογράφησης και στο διαθέσιμα κριτήρια για το θέμα των κριτηρίων πιστεύω ότι θα πρέπει να αφορούν κάθε είδους εδαφικές συνθήκες. Κάτι που ο κύριος Νίκολσον έδειξε. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, κριτήριο δηλαδή, είναι η εργασία και η εντατικότητα της εργασίας. Σε ορεινές λόγου χάρη περιοχές, αυτά σχετίζονται και με την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να μας αποσχολήσει η απόσταση από τις αγορές. ή από τις πηγές των πρώτων υλών για τους γεωργούς. Αυτά θα πρέπει να είναι από τα πρώτα κριτήρια. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Εξ ονόματος της ομάδας του, Συνοτικής Αριστεράς, το λόγο έχει ο κύριος Ενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο μας χρειάζεται τους απαραίτητους λεπτομερείς χάρτες για την υιοθετήση των μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Είναι κρίσιμο αυτό για τους εξή δύο λόγους τουλάχιστον. Πρώτος λόγος είναι θέμα σεβασμού. Το κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που έχει δημοκρατική νομιμότητα στην Ένωση και θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται για να κάνει τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Ο δεύτερος λόγος είναι θέμα κοινή λογικής σε σχέση με τις ιορικές φιλοδοξίες στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να έχουμε αλληλεγγύη με μεταξύ των εδαφών στην Ένωση. Αν θέλουμε να έχουμε αυτόνομη, αηφόρο γεωργία, με ανανεώσιμη ε, μορφή ενέργεια, με συμμετοχή στη δημόσια υγεία των καταναλωτών, με καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και που να απαντά και στι διατροφικέ ανάγκε του πληθυσμού, τότε όλε οι ευρωπαϊκέ ενισχύσει θα πρέπει να επανεξαρτηστούν με βάση αυτά τα κριτήρια και αυτού του στόχου. Και για να ε, κατευθυνθούμε προ τα εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τι λεπτομερεί χάρτε για να κάνουμε τη δουλειά μα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Μια κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί να είναι υπόθεση κερδοσκοπίας των αγορών. Είναι θέμα πολιτισμού που άπτεται όλων των πτυχών της ζωής των πολιτών των κρατών μελών μας. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Για ένα λεπτό η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπανε πολλοί σε αυτή τη συζήτηση, ε, είναι πολύ σημαντικέ οι περιοχέ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ένα νησί τι προβλήματα έχει και στην Ιρλανδία το 75% τη γη είναι ήδη σε αυτό το πρόγραμμα. Όπως και άλλοι κύριε Υπουργέ, με λυπεί το γεγονό ότι ήρθατε εδώ με τόσο ασθενεί πληροφορίες μεταξύ των, είμαστε συνομεθέτε και συμμετέχουμε στη διαδικασία της μεταρρύθμισης κοινή γεωργική πολιτική και πρέπει να σα πω ότι δεν αρκούν αυτά. Για του γεωργού στην Ιρλανδία είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τι θα συνέπειες θα υπάρχουν. Στη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέπειε θα πρέπει να υπάρχουν, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, ποιε περιοχέ θα αποκλειστούν και θέλουμε να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα περιφερειακής ευελιξίας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, και σε αυτή την περίπτωση για τις μειονεκτικές περιοχές. Θέλουμε να ξέρουμε και πότε θα εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για το 2014 και ε, πρέπει να ολοκληρωθεί ο χάρτης για τις περιοχές με τους φυσικούς περιορισμούς. Θα πρέπει όμως πριν να γίνει αυτό να εξετάσουμε όλες τις πτυχές. Ευχαριστώ. Θυμίζω ότι ένα λεπτό αποτελείται από 60 δεύτερα και έχω λόγο που το κάνω αυτό. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, σιγά σιγά θα ήταν και αστείο, θα το κάναμε και σκέτς. Αλλά λέτε ότι θα πρέπει να δηλώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο Συμβούλιο ε, λένε ε, ότι δεν ε, πρέπει να το διαβιβάσετε στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά Ποια είναι τα κράτη-μέλη και ποιο είναι το Συμβούλιο. Είναι διαφορετικά πράγματα το ένα και το άλλο και δίνουν κάποια στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι σε εμά. Τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη τι είναι. Να έχουμε του χάρτε εκείνου των κρατών μελών ε, που ε, έχουν διαβιβαστεί ε, στα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εφτασφράγιστο κοιτάπι αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζει κανεί ποιοι είναι αυτοί οι χάρτε. Ε, και είναι τίποτα πανάκριβε μετοχέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί το κάνετε έτσι. Και δεν είναι μόνο τα φυσικά ε, όρια και ε, το είδος ε, του εδάφους, αλλά και η γονιμότητα του εδάφους. Και θα πρέπει στην Ένωση να μην υπερβάλλουμε ως προς την ομιγενοποίηση γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση. Γι' αυτό πιστεύω και ζητώ να ξαναδούμε αυτό το θέμα με την ησυχία μας, αντικειμενικά, χωρίς πίεση χρόνου. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της ΚΑΠ αυτό, αλλά σε ειδική έκθεση ξεχωριστή. Και ακριβώς επειδή δεν μας πιέζει ο χρόνος και ε, ε, ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι τόσο θολή και σκοτεινή και δεν θα πρέπει να χαθεί αυτό το σημαντικό θέμα στη μεγάλη ιστορία της αναθεώρησης της ΚΑΠ και επειδή πρόκειται για μειονεκτικές περιοχές. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι οι αγρότες, οι οικογένειές τους, το εισόδημά τους και θα πρέπει με την ησυχία μας να το εξετάσουμε και να αποφασίσουμε αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε γαλάζια κάρτα του κυρίου Κούν. Τη δέχεστε την ερώτηση. βεβαίω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Γιάν, δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι το σύστημα των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών ανατρέπει το όλο εγχείρημα. Αν διάβασα σωστά, εσείς ο ίδιος ως νέος αγρότης στο Μεκλεμβούργο σε μια κρίσιμη ε, περιοχή ε, δραστηριοποιηθήκατε και ε, απεκτήσατε εμπειρία. Και είναι ακριβώς συγκεκριμένα τα σημεία, 20 σημεία για το τι συνιστά μια μειονεκτική περιοχή. Και πώς βλέπετε τις εξελίξεις και τι συνέπειες θα έχουν αυτές για τους αγρότες μας στις μειονεκτικές περιοχές. Μπορώ να απαντήσω, Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, ίσως γι' αυτό το λόγο το κρατούν κρυφό αυτό το έγγραφο και τους χάρτες, γιατί μπορούν να προκύψουν κάποια στοιχεία που δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει ούτε με την πείρα του, ούτε με την κοινωνική λογική. Από την περιοχή Άιφελ είχα επισκέπτες πριν από λίγο καιρό, που είναι ε, το ίδιο έδαφος, αντίστοιχες συνθήκες και ε, ξαφνικά η μισή περιοχή έχει εξαιρεθεί. Δεν είναι πια μειονεκτική, λέει. Μα αυτό πώ θα του εξηγήσουμε ότι ισχύει στην ευρωπαϊκή πολιτική και αφοβούνται τα κράτη-μέλη να μα δώσουν του χάρτε. Ε, τότε δεν ξέρω πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ απαιτώ διαφάνεια εδώ και ε, ειλικρίνεια. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, για ένα λεπτό, η κυρία Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και η πλειονότητα των συναδέλφων, θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω ότι απαιτείται από πλευρά Κοινοβουλίου να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε και το έργο μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ιδίω σε ένα τόσο δύσκολο πλαίσιο σαν αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για τον κλάδο επειδή δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Δεύτερον, ήδη από το Μάιο του 2010 το Κοινοβούλιο είχε εκφράσει την άποψή του για το θέμα αυτό που αφορά τις μειονεκτικές περιοχές και θεωρούμε ότι τα καθαρά βιοφυσικά κριτήρια δεν ήταν τα κατάλληλα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι να μελετηθούν και να συμπεριληφθούν και τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Διότι υπάρχουν πολλέ περιοχέ τη υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή ε, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ακριβώ λόγω τη εγκατάλειψη του πληθυσμού ε, των περιοχών αυτών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, ξεχάσουμε ότι υπάρχει και αυτό το κριτήριο και θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό και μισό ο κύριος Αλγουόρτ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, το θέμα των μειονεκτικών περιοχών είναι τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, διότι 50% τη καλλιεργήσιμη γη, τη χρησιμοποιούμενη γη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χαρακτηριστεί ω μειονεκτική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιρλανδία έχουμε περίπου το 75% τη καλλιεργήσιμη έκταση τη χώρα που έχει χαρακτηριστεί ω μειονεκτική. Το σχετικό λοιπόν πρόγραμμα θα πρέπει να προστατεύει τι περιοχέ αυτέ και τις ε, χίλιες οικογένειες γεωργών ε, της Ιρλανδίας που πλήττονται και λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων στην Ιρλανδία. Οι γεωργοί που εργάζονται σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει και περισσότερο να εργαστούν και σε συνθήκες πιο δυσχερείς. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις και ως προς το κόστος που λαμβάνουν ε, και έχουν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση στα πλαίσια του συνολικού χαρτοφυλακίου και βάσει τη αρχή τη επικορικότητα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν πλήρη ευελιξία ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια ω δι. Δηλαδή να μπορούν να καλύψουν του γεωργού του και αυτέ οι περιοχέ να μπορούν να προχωρήσουν. Θα πρέπει να υποβληθούν αμέσω οι λεπτομερεί χάρτε από τα κράτη-μέλη ώστε να καθοριστούν οι πληρωμέ προ τι διάφορε περιοχέ διότι ξέρουμε ότι μέχρι τώρα λίγα είναι τα κρατημέλη που έκαναν κάτι τέτοιο και πολλοί αρνούνται να παραδώσουν λεπτομερεί χάρτε. Η σωστή κατηγοριοποίηση των περιοχών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, εφόσον δεν είμαστε συνεπεί. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν συγκεκριμένε οδηγίε και συστάσει στα κρατημέλη ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Για ένα λεπτό, ο κύριο Χόισλινγκ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι περιφρόνηση αυτή του Κοινοβουλίου από τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Έχει έρθει η ώρα να αντιδράσουμε αντίστοιχα και να αποφασίσουμε. Μα πώς θα αποφασίσουμε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις. Περίεργο παιχνιδάκι μου φαίνεται αυτό. Ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι μυστήρια τα πράγματα. Από τη γερμανική κυβέρνηση δεν παίρνουμε χάρτες, αλλά μας δίνουν οι Γερμανοί αγρότες, η Ομοσπονδία τους. Ε, κάτι πάει στραβά. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, πιστεύω ότι στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ενιαία κριτήρια είτε είναι αυτά βιοφυσικά και αρκούν από μόνα τους, ε, τολμώ να το αμφισβητήσω πάρα πολύ σοβαρά. Χρειαζόμαστε και κοινοοικονομικά κριτήρια για να είμαστε δίκαιοι ε, στην καταγραφή μας. Αυτό απαιτεί περισσότερη δουλειά. Και δεν μπορεί κανείς να φτιάξει ένα ενιαίο χάρτη για όλη την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο ενιαίο. Γι' αυτό ε, στη Γεωργική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα να το συζητήσουμε με τρόπο ειλικρινή, διαφανή και όχι και κλεισμένων των θυρών δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοιες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για το θέμα αυτό εκ μέρους των πολλών γεωργών στα νοτιοδυτικά της ε, Αγγλίας που δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τη γεωργία στο Dartmouth στο... και σε άλλες μειονεκτικές περιοχές. Εδώ η ενεργή γεωργία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε τέτοιες περιοχές για πολλούς λόγους. Γιατί πρώτα απ' όλα εξασφαλίζει τη διαβίωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η όλη διαδικασία διαπραγμάτευση τη αναθεώρηση τη κοινή γεωργική πολιτική είναι σαν ε, δαμόκλειο σπάθη που επικαίνεται των ε, Ευρωπαίων Γεωργών. Φαίνεται ότι θέλουμε εδώ μια επιχειρηματική, έναν επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά είναι πολύ δυσχερέ να προχωρήσουμε επιτρέποντας την αβεβαιότητα να εξαπλώνεται και να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν υποχρεώσεις προς τις μειονεκτικές περιοχές. Οι γεωργοί της περιοχής με ελπίζουν στη δυνατότητα η έννοια της, βιο... δυνα... βιο... παραγωγής να ληφθεί υπόψη. Εάν θέλουμε εδώ να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας, θα πρέπει να μην απομακρυνόμαστε από τους γεωργούς. Εγώ όμως από τους εκλογείς μας το ακούω συνεχώς χρησιμοποιήστε σαφείς μεθόδους για τους υπολογισμούς, δώστε μας την απαραίτητη ενημέρωση και αφήστε τους τοπικούς φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει για την εκλογική τους περιφέρεια ώστε να πετύχουμε τους επιθυμητούς στόχους. Ευχαριστούμε. Επομένη για δύο λεπτά η κυρία Πατράου Νέβερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Εδώ η Επιτροπή θέλει μια συγκεκριμένη οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών βάσει βιολογικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Θα πρέπει λοιπόν να διατεθούν πληροφορίε για την ε, τρέχουσα διαδικασία και αυτό στα πλαίσια της γενικότερης αναθεώρησης της ε, ΚΑΠ που συζητιέται και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά είναι θεμελιώδη σημασία για να διατηρηθεί το γεωργικό πρότυπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η κοινή γεωργική πολιτική. Μιλάμε για επίπεδα βοήθεια που θα πρέπει να ανατρέχουν και στη θετική διακριτική μεταχείριση, εφόσον θέλουμε να επιτρέψουμε τη γεωργική παραγωγή σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να επιτρέψουμε τη ζωτικότητα των γεωργικών περιοχών τη υπαίθρου και να μην εγκαταλείπονται ή να μην ε, υπάρχει μετακίνηση του πληθυσμού από τι γεωργικέ περιοχέ και την υπεθροποσταστικά ε, κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιε δράσει να αντιλαμβάνονται και από τα κάτι μέλη και βεβαίω αυτό που θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε είναι λεπτομερεί χάρτε, η χαρτογράφηση, ώστε να υπάρξει και ο καθορισμό των ε, επιδοτήσεων που θα δεθούν. Όχι μόνο όμω βάσει των γεωλογικών και ε, φυσικών κριτηρίων αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών. Θα πρέπει να, λάβουν υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε των μειονεκτικών περιοχών των επιμέρους κρατών μελών. Πέραν λοιπόν των γεωργικών ε, συνθήκων όπως η απόσταση, η μορφολογία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παραγωγή. Τι είδους παραγωγή λόγω χάρη επικρατεί σε μια περιοχή. Εδώ η Επιτροπή δεν αναφέρεται στην απομόνωση ή την ε, ένταση της γεωργικής ε, καλλιέργειας την απόσταση από τις αγορές, την απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις ιδιαιτερότητε χωρών όπω η Πορτογαλία που έχει και υπηρετική χώρα μακρινή από την υπόλοιπη Ευρώπη ούτω ή άλλω, αλλά και υπερπόντιες περιοχές και διαμερίσματα όπως οι Ασόρες και η Μαδέιρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητή, ένα λεπτό, κύριο Ταπάιτζη. ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι και πρόεδρε, εγώ άρχισα τη σταδιοδρομή μου ως διπλωμάτης στην τότε Σοβιετική Ένωση. Και τότε υπήρχαν πολλά κρατικά μυστικά. Και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε τέτοια κρατικά μυστικά. σε ό,τι αφορά το ποιε περιφέρειες θεωρούνται μειονεκτικές ή όχι. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Στην πατρίδα μου, την Ουγγαρία, στο κέντρο της χώρας, μεταξύ του ποταμού Τίσα και του ποταμού Δούναβη, έχουμε μια περιοχή που ο την κατατάσσει σε ε, ημιέρημο. Είναι σχεδόν ερημική περιοχή και ε, δεν τους δίνεται ε, το καθεστώς της μειονεκτικής περιοχής, αλλά χωρίς ε, βελτιωτικά έργα και ε, αρδευτικά έργα δεν μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά κρίμα και ε, ντροπή και όνειδος που αποουσιάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Άσχουρθ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τις συνέπειες κάποιων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ταξινόμηση των μειονεκτικών περιοχών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποιες από αυτές τις περιοχές είναι από τις πιο όμορφες και τις πιο πλούσιες από πλευράς βιοποικιλότητας ε, της χώρας. Είναι όμως και από τις πιο ευάλωτες περιοχές. Και αυτές είναι οι περιοχές ε, για τις οποίες η στήριξη στην κοινή γεωργική πολιτική είναι ζωτική σημασία για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Επομένως, η σωστή εφαρμογή θα είναι ζωτική σημασία για αυτούς και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη ε, τρία σημεία. Να έχει ένα κατόφλι 50%. Επίσης, να χρησιμοποιήσει ένα ελάχιστο μέγεθος ε, διοικητικής μονάδας για να μπορεί να καθορίσει ποιες είναι οι δυνατότητες μιας γεωγετικής περιοχής και τέλος να δείξουν ένα βαθμό ευελιξίας στον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά μεονεκτήματα και τα βιοφυσικά ε, κριτήρια θα προσμετρούνται για να ταξινομηθεί η περιοχή ως μειονεκτική. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, για δύο λεπτά, ο κύριος Σιλβέστρης. Για να αποφύγουμε την απερίμωση και να διατηρήσουμε τον πλούτο των εδαφών μας, πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη στήριξη στους γεωργούς ε, χάρη στην επιπλέον ενίσχυση. Πρόκειται για μια βοήθεια η οποία θα δοθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου ε, και θα έχουν προϋπολογισμό 50% για τις μειονεκτούσες περιοχές κατηγορίας 1 ε, και θα υπάρχει και ένα μέγιστο στον αριθμό των εκταρίων. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται με τις μειονεκτικές περιοχές. Τα 8 βιοκριτήρια τα οποία προάγονται κατά πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγήσουν σε κατανοητά αποτελέσματα και δεν είναι προ όφελο ούτε των ίδιων των γεωργών αλλά ούτε και αυτών που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά. Και δεν θα μα βοηθήσουν να επιτύχουμε του στόχου που ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε. Το άρθρο 68 για την ε, συνδρομή στις μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να παραμείνει, θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένε ενισχύσεις, διότι βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή θα μειωθούν αυτές οι βοήθειες. Υπάρχουν κάποια προϊόντα όπως για παράδειγμα η ελαιοπαραγωγή στην Νότια Ιταλία και από ό,τι φαίνεται θα χάσει το 60% σε σχέση με τους ιστορικούς του τίτλους. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και για τα μνημεία και μας ενδιαφέρει και για οικολογικούς λόγους αλλά και για παραγωγικούς λόγους. Για οικολογικούς λόγους διότι το να αποφύγουμε την ενίσχυση σε αυτές τις ε, ε, παραγωγές σημαίνει ότι θα παρέμβουμε και στα αρδευτικά ε, στοιχεία και επίσης υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία ιστορικής σημασίας. Στην Απουλία και μόνο έχουμε 1.200 ε, γεωργούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά για ιστορικούς και μόνο λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την πρόταση αυτή και να λάβουμε υπόψη και άλλα κριτήρια και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σωρευτικά. Να υπάρχουν ένα σύνολο ε, φυσικών, γεωγραφικών κριτηρίων που θα βοηθήσουν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, η κυρία Κάντεμπαχ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύον, μπορώ να φανταστώ ότι δεν ήταν εύκολο για τη Δανική Προεδρία να μπει σήμερα στο ημικύκλιο. Αλλά δεν βλέπω πουθενά ελπίδα για το μέλλον ε, στη σημερινή κατάσταση που είναι πραγματικά πολύ άσχημη. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας Άτλαντας που αποτελείται μόνο από αυτά τα οχτώ κριτήρια μπορεί να βοηθήσει και να κοσμήσει τα σχολεία μας αλλά ε, όχι και την ε, ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, ούτε είναι ε, βάση για να οριοθετήσουμε ξανά τις περιοχές μας. Χρειαζόμαστε και ένα κριτήριο που να λαμβάνει υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και επίσης την Ήπεθρο θα πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ε, ε, και ένα, ως ένα χώρο που ζει κανείς και εργάζεται. Δεν μας βοηθούν τα γυμνά ψυχρά στοιχεία για τις βροχοπτώσεις και για το κλίμα και τα εδαφολογικά είναι ένας χώρος ζωής η Ήπεθρος. Φτιάξε ένα σωστό Ατλαντά που να λαμβάνει υπόψη του και αυτά τα κριτήρια, τα κοινωνικονομικά και τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε το θέμα των αντισταθμιστικών πληρωμών που συζητούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες μας στις εν λόγω περιφέρειες. Και θα ήθελα να τονίσω το εξή. Οι αντισταθμιστικέ πληρωμές είναι μια ιστορία επιτυχία τη Ευρωπαϊκή γεωργική Πολιτική. Βοήθησαν και συνεισέφεραν στι περιοχέ αυτέ να υπάρχει μια ε, σωστή γεωργία, να παραμείνουν οι αγρότε ή η βιοπικιλότητα, οι καλλιεργήσιμε εκτάσει και οι θέσει απασχόληση να διατηρηθούν στην Ήπεθρο. Ο κόσμος απέκτησε προοπτική για να παραμείνει στον τόπο του. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο με ένα θέμα τόσο ευαίσθητο έχουν αυτή τη μεταχείριση και τη συμπεριφορά. Ε, μιλάτε για 8 βιοφυσικά κριτήρια. Ας τα εξετάσουμε. Τι σημαίνει ότι δημιουργούμε νέες αδικίες που είναι χειρότερες και πιο άδικες από το σημερινό σύστημα, όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα οριοθέτησης. γίνεται χειρότερο το σύστημα. Στη Γερμανία 2,8 εκατομμύρια εκτάρια βγαίνουν και μπαίνουν 1,2 εκατομμύρια νέα εκτάρια. Όταν το συζητώ με αγρότες από τις περιφέρειες αυτές εκπλήσονται που ξαφνικά χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές περιφέρειες. Από τη Γαλλία ακούμε ότι μειονεκτική περιοχή χαρακτηρίζεται μια περιφέρεια όπου οι αγρότες έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα κατά μέσο όρο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα έχετε σκεφτεί, ε, είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε αγαπητό Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συνθήκης της Αβώνας για να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Και δεν μπορώ αστειευόμενος παρά να πω ότι να δώσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη διαβάσουν και να την εφαρμόσουν, γιατί μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί ότι ισχύει ήδη. Τα είπε και ο συνάδελφος Πέτερ Γιάρ ότι περίπου θα κάνουμε σε λίγο ε, σκέτς ε, με αυτή την ιστορία και ε, κομική παρουσίαση. Πάνω από 66% της προφορίας είναι απόρριτη και κρυφή για μας. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι διαπιστώνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είναι αποφασισμένοι να καθορίσουν πού θα βρίσκονται γεωγραφικά αυτές οι μειονεκτικές περιοχές. Αλλά αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα πόρα απέχει από το επιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι αυτές οι περιοχές ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, ε, βλέπω να εφαρμόζονται και αρκετά κριτήρια, ιδίως σε σύγκριση με τα ε, κατάλληλα σύνορα των Δήμων. Οι Δήμοι είναι διαφορετικοί από τη μία χώρα στην άλλη και στην Πολωνία. Ένας Δήμος είναι κατά μέσο όρων 12.000 εκτάρια. Και φυσικά ο κάθε Δήμος, σε κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική έκταση. Επομένως δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών Δήμων στα κράτη-μέλη. δεν θα μπορούμε να έχουμε ομογενείς περιοχές ε, και δήμους ε, που να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα και θα είναι και τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα ε, σε σχέση με αυτά που θα έχουμε σε μια άλλη χώρα. Και διαπιστώνουμε ότι το 66% το οποίο θα αποτελέσει το κατόφλι για να ξεκινήσουν οι ενισχύσεις, είναι πάρα πολύ υψηλό, διότι οι περισσότερες περιοχές θα είναι εκτός αυτού του ορισμού και επομένως οι γεωργοί δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν πλέον. Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις στην Πολωνία ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει σοβιά οποιασδήποτε μορφέ, αν δεν υπάρχει κατάλληλη ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ που ζητούν αυθόρμητα το λόγο οι συνάδελφοι. Για ένα λεπτό, κύριο Φερχέιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο Συμβούλιο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς δεν εκπροσωπείται με τον τρόπο που θα επιθυμούσα λόγω σεβασμού από το Κοινοβούλιο. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια που λέγεται Άιφελ στη Γερμανία και πλήττεται τρομακτικά από τα νέα μέτρα. Και διαρωτώ με, γιατί αυτά τα κριτήρια ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των περιοχών αυτών δεν έχουμε και τι απαραίτητε προφορίες για να αποφασίσουμε με τα λόγου γνώσεως. Και έχει γίνει μια μελέτη αντικτύπου σοβαρή και σωστή για να αντιποκριθούμε στους αγρότες δεν αρκούν τα βιοφυσικά κριτήρια, χρειάζονται οπωσδήποτε και κοινωνικο-οικονομικά. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το σημαντικό στοιχείο να το εξετάσει με την ησυχία της ξεχωριστά από το γενικό πακέτο της αναρρύθμισης της ΚΑΠ και μάλιστα με τα ε, απαραίτητα στοιχεία και τεκμηριωμένα για να ξανασκεφτούν τα κριτήρια και να τα ξανασυζητήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πρέντεργαστ. Um, Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πρέπει να δούμε και την, ε, το ποσοστό προχώπτωσης στα εδάφη ως ένα από τα κριτήρια που θα επιτρέψουν την επιλογή των μειονεκτικών περιοχών. Όπω το Λέμερικ στην Ιρλανδία λόγω χάρη, λόγω των ακραίων κλιματικών συνθήκων και τη ψύχρανσης του εδάφου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν λεπτομερεί χάρτε για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη δική σα την απόκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν λάβαμε διευκρινήσει από το Συμβούλιο, αλλά αρκετά είναι τα κράτη-μέλη που έχουν πληροφορίες και τελικά δεν απέστειλαν τα στοιχεία τους. Από ό,τι κατάλαβα, 20 κράτη-μέλη διαθέτουν πληροφορίες και 12 μπορούν να τις παρουσιάσουν εδώ και στην αίθουσα. Κάποιοι άλλοι είναι σαν να έχουν ανακαλύψει χρυσό και να μην θέλουν να μα δώσουν αυτή τη σημαντική είδηση. Όμω μιλάμε για ένα ζήτημα πολύ πολιτικά ευαίσθητο. Θα πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουν όλοι και οι υπεύθυνοι τη Επιτροπή που έχουν χαρακτηρίσει τι μειονεκτικέ περιοχέ. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσει και σε σχέση με την αναθεώρηση τη κοινή γεωργική πολιτική αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα έλεγα λοιπόν στο Συμβούλιο να μην λέει στο Συμβούλιο να αποταθεί στην Επιτροπή για να ζητήσει τις πληροφορίες, αλλά να συνεργαστούμε, να γίνουμε ένα στην προσπάθεια αυτή να απαιτήσουμε πληροφορίες από όσους δεν τις έχουν παράσχει. Άκουσα συναδέλφους και από άλλα κρατημέλη να λένε το ίδιο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν εδώ. Οι πληρωμές αυτές είναι καθοριστικές για την επιβίωση των γεωργών στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα έλεγα λοιπόν πριν θέσουμε ερωτήματα προς εμάς τους ιδίους να αναρωτηθείτε εσείς τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ κύριε Μάνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ε, μειονεκτικές περιοχές είναι πολύ σημαντικές για τη γεωργία μας αν θέλουμε να διατηρήσουμε παντού γεωργική παραγωγή και είναι και σημαντικό αυτό για την ασφάλεια και την επιστημιστική. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη δεν επικρατούν οι ίδιες μετρολογικές συνθήκες. Εγώ είμαι Φιλανδή. Ε, το χειμώνα έχουμε πολύ χιόνι και ακόμα και τώρα που είναι Απρίλιος έχουμε ένα μέτρο χιόνι. Δηλαδή, αυτά τα βιοφυσικά κριτήρια θα πρέπει να είναι μεν τα πρώτα κριτήρια που λαμβάνει κανείς υπόψη του στον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών. Τι γίνεται με το κλίμα, ε, αν είναι πολύ βαρύ το ψύχο στο χειμώνα και πολύ σύντομη η περίοδος ε, ανάπτυξης ε, των φυτών και πολύ μικρή η περίοδος μέχρι τη θα πρέπει όλα αυτά να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέα έχει το λόγο που είχε προηγουμένως κανονικά λόγω χρονογόρευσης, αλλά δεν ήταν παρόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ο συντάκτης της ερώτησης αυτής θα χρειαζόμουν δύο λεπτά. Πόσο χρόνο έχω για αυτή την παρέμβαση, λοιπόν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να γίνει εδώ μια απαραίτητη διευκρίνηση για την όλη συζήτηση. Η κατηγοριοποίηση των μειονεκτικών περιοχών του 2005 με περιβαλλοντικά και κοινωνικονομικά κριτήρια έχει πλήξει κάποιε από τι πιο μειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μικρή κλίμακα γεωργία και η οικογενειακή κλίμακα γεωργίας έχουν πληγεί ιδιαίτερω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αρνείται εδώ να μας δώσει το ρόλο που πρέπει να αναλάβουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινή γεωργικής πολιτικής και ουσιαστικά δεν μα επιτρέπει να προστατεύσουμε τι μειονεκτέ περιοχέ. Υπάρχουν βεβαίω τα κριτήρια, τα γεωλογικά, τα μορφολογικά, τα περιβαλλοντικά πρέπει να υπόψη, αλλά κυρίω τα οικονομικά και οικονομικά, γιατί υπάρχουν αδικίε και ανισότητε εδώ. Για την κατανομή των κονδυλίων ε, τη κοινή γεωλογική πολιτική μεταξύ κατομελών και γεωργών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να διευρύνουμε τα κριτήρια και να τα διαφοροποιήσουμε, ιδίω τα κοινωνικο-οικονομικά. Ω προ του δείκτε απερίμωση, λόγου χάρη τη ε, υπαίθρου και τη κάλυψη τη υπαίθρου. Εδώ λοιπόν για τα περιβαλλοντικά κριτήρια έχει αναθέσει σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητα να τα καθορίσουν. Όμω εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν πρόσωποι και από τα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό δεν έγινε και μία ερώτηση που σας απίφθηνα το 2010 μας δείχνει ότι σε καμία περίπτωση Πορτογάλος εμπειρογνώμων δεν συμμετείχε σε αυτή την ομάδα. Και αυτό έγινε με τη συντηρητική πλειοψηφία των κρατών μελών. Οι εμπειρογνώμονε είναι γνωστοί, Όμω, πέραν των διαφορετικών καταστάσεων που ισχύουν σε κάθε κράτο μέλο, είναι δύσκολο να βρούμε εναρμονισμένα κριτήρια με τόσα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι, Κάποιοι ωφελούνται ει βάρο άλλων, όπω συνήθω συμβαίνει. Λοιπόν, στα πλαίσια τη κοινή γεωργική πολιτική, ένα θεμελίδιο ερώτημα παραμένει χωρί απάντηση. Πώ θα εγγυηθούμε τη δίκαιη κατανομή των κονδυλίων τη κοινή γεωργική πολιτική, πώ σε κάθε εκατό μέλο θα εγγυηθούμε το δικαίωμα παραγωγή και επισητιστική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις μόνο, γιατί έχω καλυφθεί από τους συναδέλφους. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί απουσία σαφών ορισμών ως προς τις μειονεκτικές περιοχές. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση στις προσωμιώσεις. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε κάτι το οποίο αγνοούμε. Το Κοινοβούλιο καλείται να εξηγήσει στους πολίτες τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με αδιαφάνεια ε, θα είναι αθέμητη και παράνομη και θα ε, προσβληθεί. Επίση, θα πρέπει να καταλάβει το Συμβούλιο ότι έχει λόγο και το Κοινοβούλιο. Οι αγρότες περιμένουν ε, να ε, συμπεριλαμβάνονται όλα τα κριτήρια και τα γεωγραφικά και τα κοινωνικο-οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη εκπρόσωπη του Συμβουλίου. Σήμερα ακούσαμε τη θέση σας και νομίζω ότι αποτελεί πραγματικά προσβολή προς το Κοινοβούλιο είναι προσβολή προς το Κοινοβούλιο, διότι δεν μας θεωρείται επίσης όρις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, τα οποία ε, νομοθετούν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και εγώ ως εισηγητής της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής δεν το δέχομαι, να αποφασίσουμε και να προτείνουμε τη θέση μας χωρίς να γνωρίζουμε και χωρίς να διαθέτουμε τις ίδιες πληροφορίες που διαθέτετε και εσείς τις επιπτώσεις για τον πρώτο πυλώνα και τις ε, άμεσες ενισχύσεις της ποσόστοσης η οποία θα δοθεί για τις μειονεκτικές περιοχές ε, τις οποίες δεν μπορούμε να προσωμιώσουμε εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα δεδομένα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να σας δώσει απάντηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής εάν δεν μας διαθέσετε τα απαραίτητα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ποιος ζήτησε το λόγο. Κύριε Σφέρ. Ε, πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εγώ είμαι Σλοβένος. Για τη χώρα μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσωμιώσεις. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και να πω ότι τα βιοφυσικά κριτήρια δεν αρκούν για να ορίσουμε τις περιοχές αυτές. Είναι και τα κοινωνικο-οικονομικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα όμως να τονίσω κάτι που δεν υπόθηκε ακόμα σήμερα. Υπάρχει και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη στην Ήπεθρο. Οι νέοι αγρότες είναι πάρα πολύ λίγοι και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Πριν από λίγες μέρες στο Κοινοβούλιο έκανα αντίστοιχη ακρόαση και διαπιστώθηκε ότι μόλις το 6% των ε, νέων απασχολούνται στη Γεωργία, μάλιστα ε, νέοι ηλικία κάτω των 35 ετών. Και αυτό το κριτήριο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την υπόδειξή σας ad hoc. Θέλει κανείς άλλο το λόγο στο Κατσιέ. Ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Κέλλη, πείτε. Δεν είχα σκοπό να λάβω το λόγο. Ήθελα περισσότερο να ακούσω τι είχατε να πείτε, αλλά πρέπει να πω ότι πλέχτηκα με τη συζήτηση και θα ήθελα να ακούσω κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσει. Καταρχά, ο κύριος Νίκολσον αναφέρθηκε στο ελεκτικό συνέδριο και είπε ότι θα μπορούσε ίσως να ε, εξηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια επιπλέον επ' αυτού. Και δεύτερον, για αυτή τη νέα ταξινόμηση. Ο κύριος Ντές μας είπε ότι η Γερμανία θα χάσει κάποιες περιοχές ε, και στο στόχο 2. Ουσιαστικά είναι σαν να μετακινούμε μια πινέζα και να αλλάζουμε τις ε, γεωγραφικές κατανομές και τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακούσαμε. Ε, κάτι είναι σάπιο εδώ και θα πρέπει πραγματικά να ακούσουμε την απάντηση για να δούμε τι γίνεται και με την κοινή γεωργική ε, ε, πολιτική και προ όφελο γενικότερα τη πολιτική και των Ιρλανδών πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Προ το παρόν δεν ζητεί κανεί άλλο το λόγο στο ΚΑΤΖΙΑΙ. Θα παρακαλέσω τον Προεδρεύοντα να λάβει το λόγο για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι λένε ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια για το θέμα αυτό και λαμβάνονται αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών. Και όπως σας είπα και στην αρχή της παρέμβασής μας, Ζητήσαμε περισσότερα στοιχεία και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να ξανασκεφτούν τη θέση τους ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ε, και έγκυσε να συζητήσουμε τα θέματα που συζητούσαμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε διαφάνεια και από πλευράς Προεδρίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει διαφάνεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις θέσεις που εκφράσετε και για τη συζήτηση. Ε, Εγώ σας ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, Θα να σας ε, ε, ενημερώσω ότι